Συνεχίζεται η συνεδρίαση. Ξαναρχίζει η συνεδρίαση. Θα σα διαβάσω το αποτέλεσμα των εκλογών σε λίγα λεπτά. Θα ήθελα να σα πω τι έγινε στο δεύτερο γύρο. 660 ψήφοι. Έδωσαν 11 άκυροι, 649 έγκυροι ψήφοι. 725 θα ήταν, είναι η απόλυτη πλειοψηφία. Οι υποψήφοι έχουν τους εξής ε, ψήφους. 266 για την Ρομπέρτα Αντζελίνη. 259 Ιζαμπέλ Ντουρόν. 175 Μιχάλ Καμίνσκι. 141 Σιλβάνα Κοχμαρίν Μερίν. 242 Μακμίλαν Σκότ. 292 ε, Ματίνε Ματίνε. 288 Νταγμαρότ Μέρτα 276 Λίμπο Ρούτσεκ 239 Παλ Σμιτ 303 Ελέχο Βιδάλ Κφάτρας 274 Ταϊάννα Βόλη. <coughs> και 235 Ράινα Βίλαντ Jeśli chodzi o kandydatów, którzy otrzymali bezwzględną większość oddanych głosów, οι υποψήφοι που είχαν την απόλυτη πλειοψηφία είναι οι εξή. Κανεί. Κανένα δεν πέτυχε την απόλυτη πλειοψηφία που απαιτεί το. Παραμένουν λοιπόν 11 έντρε αντιπροέδρων που πρέπει να πληρωθούν. Σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει να έχουμε ένα τρίτο γύρο εκλογών. Εάν δεν διαφωνεί κανένας, θεωρώ ότι θα παραμείνουμε με τον ίδιο κατάλογο των υποψηφίων. Ε, δεν βλέπω να διαφωνεί κανείς.